Καλή σας ημέρα. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Στόχος του πρώτου μερού της σημερινή συνεδρίασης είναι η εκλογή του Προέδρου και των τεσσάρων αντιπροέδρων. Θα περάσω τώρα στην εκλογή του Προέδρου μας. Μήπως υπάρχουν προτάσεις από πλευράς πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γκάλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω τον προηγούμενο τον συνάδελφό μας Ανών Ντανζό. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ. Αν υπάρχει μόνο ένα ε, υποψήφιος, σε διαβοή εκλέγεται ο πρόεδρος. Μπορείτε να περάσετε παρακαλώ και να καταλάβετε τη δέκα. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η δυνατότητα να αναλάβω την Προεδρία στην Υποεπιτροπή αυτή που ελπίζω ελπίζω να αναπτύξει τις εργασίες σας σύμφωνα με όσα προτείναμε πρόσφατα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Πιστεύω ότι είναι ένας σωστός δρόμος που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε πολύ περισσότερο από ό,τι κάναμε ως τώρα θέτοντας μία διπλή προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που έχουμε αναπτύξει στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι το πρώτο στο καθήκον μας, και δεύτερον σε ό,τι αφορά το δυναμικό μας, κάτι που έγινε μέσω των εργασιών που βασίστηκα στην έκθεση του πρώτου αντιπροέδρου του Κριστόφ Λιζέκα που υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο Στρασβούργο. Και πιστεύω ότι ανοίγει το δρόμο για μια συνέχεια που θα πρέπει να είναι η ιδιαίτερα αποτελεσματική από μέρους μας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με επικοδομητικό τρόπο όπως κάναμε ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Περνάμε τώρα στην εκλογή των αντιπροέδρων. Ξεκινάμε με την εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Ποιες είναι οι προτάσεις, παρακαλώ, από πλευρά των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Η πρότασή μου αφορά το συνάδελφο Μαυρονικόλα. Merci. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαυρονικόλα. Ε, υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Κύριε Μαυρονικόλα, δέχεστε την πρόταση αυτή, την υποψηφιότητα. Κύριε Μαυρονικόλα, ο κύριος Μαυρονικόλας ελέγχεται πρώτο, ε, ε πρώτος αντιπρόεδρος. Συνεχίζουμε με την εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου. Μας έχει να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις των πολιτικών ομάδων. ενημερωθήκαμε από την ομάδα Αντέλ. Κυρία Νικολάη προτείνεται. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες όχι η κυρία Νικολάη. Συνεπώς εκλέγεται ως δεύτερη αντιπρόεδρος. κυρία Νικολάη δεν είναι παρούσα. Εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου πρόταση των πολιτικών ομάδων. Εγώ προτείνω τον κύριο Παλέτα. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Ο κύριος Παλέσκης δέχεται. Ωραία, ο κύριος Παλέσκη εκλέγεται τρίτος αντιπρόεδρος τη Επιτροπής, μα. Επιτροπής μας. Τέταρτος αντιπρόεδρος, πρώτες στο πολιτικό ομάδο, ο κύριος Γκαλέρ. Προτείνω τον Κριστόφ Λιζέκ στη θέση του τετάρτου αντιπροέδρου. Εάν δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις, ο κύριος Λιζέκ συμφωνεί, συνεπώς εκλέγεται τέταρτος αντιπρόεδρος. Θερμά συγχαρητήρια. Όπως διαπιστώνεται η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας χαρακτηρίζεται από μεγάλη σταθερότητα κάτι που αποτελεί καλό ιονό. Θα σας παρακαλούσα να διακόψουμε για λίγα λεπτά για να τακτοποιηθούν ε, οι καλεσμένοι μας και μετά θα ξεκινήσουμε κανονικά τη συνεδρίασή μας, την οποία θα την αφιερώσουμε στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε δύο λεπτά ξεκινάμε και πάλι. Euh, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε και πάλι τις εργασίες μας. Θα ήθελα να σας ε, δώσω ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία για το τομέα δράσης μας. Στις 15 Δεκεμβρίου η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε με βάση διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του διευρυμένου Προεδρίου της Υποεπιτροπής και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να δραστηριοποιήσει την Υποεπιτροπή μας και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκ παραλίλου. Συνεπώς συμφωνήθηκε ότι η Υποεπιτροπή μας θα μπορούσε να συντάξει δύο προτάσεις ε, πρωτοβουλίας αντί για... Τρει. Τρεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν εκ παραλίλου να συντάξουμε τρεις εκθέσεις, κάτι που συζητήσαμε, θα συζητήσουμε στην ομάδα του Προεδρείου που θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντί για 8 έχουμε 12 εμπειρογνώμονες, αυξήθηκε ο αριθμός του και έχουμε και κάτι αντίστοιχο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και αυτό αφορά το προπολογισμό των εμπειρογνωμών. Ο εσωτερικός κανονισμός είναι υπό αναθεώρηση για να μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτές τις αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και να διευρύνουμε το πεδίο δράσης μας. Στις 23 Ιανουαρίου 2012, δηλαδή πριν από δύο μέρες, ενδεχομένω το διαβάσατε, το Συμβούλιο διόρισε τον στρατηγό Πατήκ Τερουζιέ, πρόεδρο ε, σε αντικατάσταση του στρατηγού Σιρένα, ο στρατηγός Αντερουζιέ θα αναλάβει στο τέλος του χρόνου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον προσκαλέσουμε στην υποεπιτροπή μας. Σήμερα το απόγευμα θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Αποκινούμε την ΑΦΕΤ θα δεχτούμε τον ειδικό εντεταλμένο που έχει οριστεί για το κέρας της Αφρικής, τον κύριο Ραντός, που φαντάζομαι ότι όλοι σας γνωρίζετε. Καλώς ορίσατε κύριε Στίβενς, κύριε Πρέσβη. Το προηγούμενο Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης, θίξαμε το θέμα των προτάσεων που είχαν υποβληθεί από την ομάδα της Βαϊμάρης Πλάς, Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία έτσι ώστε η, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα είχε τη δυνατότητα προγραμματισμού για τις διάφορες στρατιωτικές δράσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα ήταν ιδιαίτερα ζωντανή. Δεν μπόρεσε να επιτευχθεί μια συμφωνία το Συμβούλιο όμως εξέφρασε τη συμφωνία του για να ε, αναπτύξει δράσεις το κέντρο ε, επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορέσει να προγραμματιστεί μια νέα αποστολή που είναι υπό προπαρασκευή και που αφορά την ενίσχυση ε, των δυνάμεων στον κέρας της Αφρικής. Η ενεργοποίηση του κέντρου επιχειρήσεων υπόκειται σε μια νέα απόφαση του Συμβουλίου για να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, γιατί επικρατεί μια κάποια σύγχυση θα λέγαμε, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο ε, ο Διευθυντής ε, της ε, M5, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού, να μας δώσει ορισμένες διευκρινήσεις. Θα ενημερωθούμε και για την προετοιμασία της νέας αυτής επιχείρησης και για το συντονισμό με δύο άλλες επιχειρήσεις στην ε, στο κέρας Αφρικής, ε, στην ε, Ταϊλάνδη και στη Σομαλία και αυτό σημαίνει ότι το κέρας της Αφρικής γίνεται ένα προσκήνιο επιχειρήσεων ιδιαίτερα σημαντικό. Ένα κέντρο επιχειρήσεων θεωρητικό, γιατί δεν είμαστε όλοι μας εξοικειωμένοι με αυτή τη δομή που δίχως άλλο θα καταλάβουμε κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Θα καταλάβουμε και ορισμένα πρακτικά θέματα. Ο κύριο Στίβενς καταρχάς από πλευράς ε, της Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ που μας καλέσατε για να κάνουμε αυτές τις διευκρινήσεις και να έχουμε αυτή τη συζήτηση εδώ ενώπιόν σας. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ και θα μου το επιτρέψετε αυτό για την εκλογή σας καθώς επίσης και όλους τους αντιπροέδρους για τη εκλογή τους. Επιτρέψτε μου επίσης και για άλλα ευτυχή γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην προσωπική σας ζωή. Θέλω να συγχαρώ και γι' αυτό. Ε, για την την ενεργοποίηση του... Ξεκίνησε το Δεκέμβριο το Συμβούλιο, ξέρω πως γνωρίζετε πάρα πολύ, ο οποίος ε, αποτελείται από τους υπουργούς... είπε ότι θα ενεργοποιήσει αυτό το κέντρο λειτουργίας με τις δυνατότητες οι οποίες έχουν να ποιού Και βεβαίως αυτό το πρέπει να στα συμπεράσματα. Για να... Για να υπάρχει μια επιτάχυση αυτής της ενεργοποίησης όσον αφορά το κέρας τη Αφρικής, έτσι, στις 6 Δεκεμβρίου ξεκίνησε σε αυτό το κείμενο επιχειρήσεων ένα κείμενο το οποίο προέκυψε και, και είναι πάρα πολύ γνωστό ε, σημαντικό να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς πώς μπορεί να γίνει αυτή η, επιτύχη, η επιτάχυση, πώς μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ διαφόρων αποστολών που γίνεται στο κέρας της Αφρικής εναντίον της ε, πειρατείας, καθώς επίσης και το δυνάμενο κοινό οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν, καθώς επίσης και μια νέα αποστολή η οποία βασίζεται σε, η οποία είναι βέβαια πολιτικής μορφής αλλά βέβαια έχει και μια στήριξη στρατιωτική. Έχουν απτύξει λοιπόν όλα αυτά και αυτά παρουσιάστηκαν στο PSE, στο κέντρο επιχειρήσεων για περαιτέρω διευκρινήσεις και εξέταση. Επίσης, το κέντρο αυτό, στο κέντρο αυτό έγιναν πολλές συζητήσεις όσον αφορά αυτή στις 18 18-19 Ιανουαρίου γιατί καθώς επίσης δόθηκαν γνωμοδοτήσεις στρατιωτικού περιεχομένου και με βάση όλα αυτά είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε αυτό το κέντρο επιχειρήσεων για πρώτη φορά από τη στιγμή εκείνη που δημιουργήθηκε σαν μια δυνατότητα που δίνεται σε ένα κέντρο όταν δημιουργήθηκε λοιπόν το 2004. Το έχετε δει ήδη αυτή τη στιγμή και το έχετε να ότι το Συμβούλιο την τελευταία Δευτέρα έδωσε την τελική μορφή την συμπολιτική συμφωνία που υπήρξε για την εργοποίηση καθώς επίσης και τα συμπεράσματα, τα πορίσματα τα οποία υπάρχουν σε πολιτικό επίπεδο Μερικές χώρες βεβαίως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περάσουν αυτό το κείμενο διαμέσου του κοινοβουλευτικού ελέγχου και να εγκριθούν καθώς επίσης και οι περισσότερες λεπτομέρειες για την για τη δραστηριοποίηση του θα πρέπει να γίνει μέσα από μία απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών. Αυτό αναφέρεται βέβαια στα συμπεράσματα και ε, βεβαίως δεν έχει περατωθεί εντελώς γιατί είναι σε ένα στάδιο τελικής απόφασης. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία η οποία συνεχίζεται και η οποία μπαίνει στην τελική τη φάση και θα υπάρξει μια απόφαση του Συμβουλίου με βάση τα απορίσματα αυτού του κέντρου επιχειρήσεων καθώς επίσης και των αποφάσιο της προηγούμενης Δευτέρας του Συμβουλίου, όλα αυτά μαζί και τις αποφάσεις του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου, όπου εκεί αναφέρεται ότι το σχέδιο για τη διαστηριοποίηση, ενεργοποίηση του κέντρου επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται πριν από το επόμενο Συμβούλιο που θα γίνει ε, πριν από το επόμενο συμβούλιο που θα γινει πρωτη πρώτης 321η Ιανουαρίου τρέχοντος, ενεστώτος συγγνώμη. Ξέρετε διάφορες χώρες λοιπόν μέλη θέλουν μια επικοδομητική, μια πραγματική, ρεαλιστική προσέγγιση όλων αυτών των πραγμάτων. Γι' αυτό το θεσμικό όργανο το οποίο θα υπάρξει και κατά αυτόν τον τρόπο και μπορεί αυτό να γίνει εφόσον αποφαστεί εντάχει με μεγάλη σπουδή και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να έρθουν και να συνεπάρξουν πολιτικοί και στρατιωτικοί για να γίνει περαιτέρω συνεργασία. Βεβαίως, αυτό θα έχει μια άμεση υποστήριξη από τον επιχειρησιακό διοικητή ο οποίο θα είναι και ο αρχηγό αυτής της όλης αποστολής και οι αποστολέ του θα είναι για την καταπολέμηση της πειρατεία στη θάλασσα, ένα άλλο θα είναι για τη Σομαλία και βεβαίω εκεί θα γίνει μια κατάρτιση και μια εκπαίδευση των στρατιωτικών της Σομαλίας οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν του κινδύνου που ελοχεύουν σε αυτή τη χώρα και θα υπάρξει και ένα τρίτο το οποίο θα είναι πραγματικά για οποιαδήποτε άλλη εργασία και η οποία άπτεται των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίω όπω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά υπήρχε μεγάλη επιτυχία σε αυτήν την προσπάθεια. Τώρα ξεκινήσαμε μια νέα βάση για μια νέα αποστολή η οποία θα βοηθήσει όλες εκείνες τις χώρες του κέρδου της Αφρικής για να έχουν τη δυνατότητα να υπεραμηθούν των συμφερόντων και των χωρών τους καθώς επίσης και θα βοηθήσουν το στη Σομαλία και του, το λαό της Σομαλίας για να υπάρξει μια δυνατότητα προστασίας ορισμένων ζωνών. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι είναι μια πολιτική αποστολή, μη στρατιωτική αποστολή αν θέλετε, και η οποία μπορεί να βοηθήσει τα μάλα, καθώς επίσης να υπάρξει μια καλύτερη πολιτική εμπειρογνωμοσύνη. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και υπό το φως των προσφάτων ε, αποφάσεων που έχουν όλα αυτά διευκολύνουν πάρα πολύ την κατάσταση και καλούν πραγματικά τις διάφορες χώρες να κάνουν διάφορες συνεργασίες μεταξύ τους, να υπάρξει μια συνέργεια μεταξύ των διαφόρων χωρών. Αυτό το επιχειρήσεων υποστηρίζει τις υπάρξεις δομές Επίσης το προσωπικό, το στρατιωτικό, το οποίο θα υπάρξει εκεί πέρα και θα υπάρχει μια διασύνδεση που θα υπάρχει με την Καλάστα, η οποία θα είναι σε αυτό το op center, στο κέντρο επιχειρήσεων, και θα υπάρξουν στοιχεία στήριξη, υποστήριξη, οι οποίε στρατιωτικά και μη στρατιωτικό. Όλο αυτό το σύμπλεγμα θα είναι μέσα σε αυτό το κέντρο και βεβαίω θα δίνουμε και τι λεπτομέρειε που χρειάζονται για όλε αυτέ τι αποστολέ που γίνονται και θα καλύπτει αν θέλετε όλο αυτό το χώρο με μια πληροφόρηση αν και ήθελ. Αυτό λοιπόν το κέντρο θα εξασφαλίσει την, τη λειτουργία, την αυτόνομη λειτουργία του, καθώς επίσης και τον συντονισμό που θα πρέπει να υπάρχει. Το βλέπετε αυτό ότι υπάρχει μέσα στην πρώτη απόφαση που έχετε χείρας, στο σχέδιο αυτό αποφάσεως, κεφαλή, ο ηγέτης θα διοριστεί, θα ονομαστεί εκ μέρους του Συμβουλίου των Υπουργών και βεβαίως θα είναι ένας από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την διάρκεια, τα κράτη-μέλη όπως ξέρετε είναι θέμα το οποίο υποσυζήτησαν ακόμη. Τα κράτη-μέλη συμφωνούν, συμφώνησαν, εφόσον η διαστηροποίηση βεβαίως και η ενεργοποίηση συνθέεται έχει σχέση με τη διάρκεια που θα έχει. Βεβαίως τα δύο αυτά θέματα είναι ελέγχοντα. Και το θέμα αυτό λοιπόν είναι συζήτηση πόσο διάρκεια. Γιατί μερικοί λένε ότι θα πρέπει να το επανεξετάζουμε κανονικά για να δούμε πόσο διάστημα χρόνου θα δώσουμε και, και αυτό είναι κάπως καινοτόμο θέλετε, είναι κάτι καινούριο το οποίο προκύπτει, αλλά άλλα χώρες λένε θα υπάρξει μια απόφαση εκ μέρου Συμβουλίου, εφόσον δοθεί μια πρώτη προθεσμία ενό άτσου Φερρυπίν, α πούμε, μετά θα δοθεί μια παράταση και Βέβαια αυτό πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων κατά πώ θα είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια και ούτω καθεξή για τη συνέχιση αυτή τη αποστολή. Όλα αυτά είναι βεβαίω όπω σα είπα και στην αρχή υπό συζήτηση και υπό εξέλιξη. Έτσι λοιπόν η περιοδική αντιμετώπιση, θεώρηση αυτών των πραγμάτων και η επανεξέταση είναι πάρα πολύ καλά. Έξι μήνε είναι επίσημη, μια προθεσμία είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό το κέντρο πιστεύουμε πω ξεκινάει καλά, τα πράγματα πάνε στο σωστό δρόμο και κάθε έξι μήνε θα πρέπει να υπάρχει αυτή, αυτός ο έλεγχος αν θέλετε και, και αυτή η ηγεσία η οποία θα πρέπει να υπάρχει ε, θα πρέπει να ασχολείται και με την ηγεσία αλλά και το όλο κέντρο πώς θα πρέπει να διαρθωθεί και πώς θα πρέπει να προχωράει. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση η οποία έχει ακολουθηθεί. Όσον αφορά το δημοσιονομικό τώρα καθεστώς ψάχνουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα μέσα, τα οικονομικά εννοείται βεβαίω πάντοτε, πώς ακριβώς αυτά τα κονδύλια θα τεθούν σε λειτουργία, το προσωπικό θα πρέπει να είναι ε, από το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο βρίσκεται ήδη, οι οποίοι βεβαίως έχουν και την κατάλληλη ε, εμπειρία σαν στρατιωτικοί και βεβαίως αυτό θα μπορεί να έρχεται από τα διάφορα επιτελεία των κρατών μελών και να εφαρμόσουν αυτά τα οποία έχουν αποφασίσει στο επίπεδο αυτού του υπηρεσίου κέντρου. Όλα αυτά είναι πολύ σαφή, διότι υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία στηρίζουν. Υπάρχει αυτό το liaison, αυτή η διασύνδεση η οποία γίνεται αυτό το κέντρο liaison και μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ περισσότερο την εμπειρία την οποία έχουμε. Έτσι λοιπόν το προσωπικό θα έρθει από το επιτελείο μπορεί να ε, επανδρώσει αυτό το κέντρο και τα πρόσθετα, το πρώτο κόστος θα έρθει, θα έρθει από τον προϋπολογισμό ο οποίος προβλέπει αντίστοιχα κονδύλια στις διάφορες χώρες. Είναι σαφές λοιπόν πάρα πολύ σαφές ότι στο χρηματοδότηση χρειαζόμαστε ακόμη να εργαστούμε για να υπάρχει μια βιώσιμη κατάσταση και θα πρέπει να υπάρχει πιο ρεαλιστική, πιο πραγματική για να υπάρξει καλύτερη ενεργοποίηση αυτού του κέντρου. Είναι παραπαραίτητο αυτό να γίνει, αλλά στο μέλλον πιστεύουμε ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ένα μπορούν να τεθούν κατά τέτοιο τρόπο σε εφαρμογή, ούτω ώστε να υπάρξει ένα βιώσιμο τρόπο ε, επιβίωση αυτού του κέντρου, εφόσον θα παραστεί ανάγκη να λειτουργήσει πέρα ενό ή δύο ετών. Θα ήθελα πρώτα να σταματήσω εδώ. Ε, φρονώ πω οι συστάσει τι οποίε έχουμε κάνει για αυτό το επιχειρησιακό κέντρο και έρχονται στοιχεία τα οποία στηρίζουν τη διάθεση την οποία υπήρξε όσον αφορά τις αποστελές τις οποίες θα πρέπει να επιτελέσει αυτό και πιστεύουμε ότι υπάρχουν στις δομές είναι τέτοιες οι οποίες βοηθούν περισσότερο αυτές οι δομές σε μια αύξηση, επάυξηση της συνεργασίας, καθώς επίσης και μια καλύτερη συνέργεια την οποία μπορεί να υπάρχει με διαφόρων χωρών σε αυτό το θέμα, για την επιτυχία των αποστολών, οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια αυτού του επιχειρησιακού συγγνώμη, κέντρου και και νομίζω πως πραγματικά θα λειτουργήσει με έναν αποτελεσματικό τρόπο εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν περάσουμε ε, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, υπάρχουν μέσα ερωτήσει οι οποίε ετέθησε. Ο κ. Γκάλερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Στίβενς. Ε, θα ήθελα καταρχάς να διαπιστώσω πολιτικά ότι χαίρομαι ειδικότερα που έχουμε δείξει το θέμα του επιχειρησιακού κέντρου από το ακρόνιμο OSQ ε, πήγαμε στο OSC. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συντονισμό, είναι ξεκάθαρο αυτό και γι' αυτό ε, χαίρομαι ιδιαίτερως ε, για τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Όσον αφορά στην διάρκεια της ενεργοποίησης. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι αν θέλουμε να περιοριστεί σε ένα χρόνο, η Μεγάλη Βρετανία δεν θέλει να γίνει κάτι τέτοιο για παράδειγμα, ίσως θα πρέπει να μας πείτε ε, από πού προέρχονται οι δισταγμοί του Κοινοβουλίου, γιατί από τη Μεγάλη Βρετανία δεν προέρχονται. Ε, με ενδιαφέρει να μάθω από πού προέρχονται. Επιπλέον, αναρωτιέμαι εάν έχει κάποιο νόημα ο σχεδιασμός, γιατί διαβάζω εδώ στα συμπεράσματα ότι το κέντρο επιχειρήσεων μεταξύ άλλων θα δίνει υποστήριξη στον ε, διοικητή για τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα δεν θα είναι μόνο ένα ε, στρατηγείο στρατιωτικό, αλλά θα έχει και μη στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις ε, που θα στηρίζονται από τον ε, διοικητή. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς έχουν τα πράγματα στη συζήτηση αυτή και τελικά πολιτικά να ξέρουμε πώς ε, θα πρέπει να αντιδράσουμε όταν υπάρχουν ε, ε, αντιδράσεις διοικητικές, ας πούμε. Ο κύριος Γκόλτ Τιερή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εννοείται ότι εμείς είμαστε υπέρ οποιοδήποτε βήματος γίνεται σε αυτόν τον τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να αυξηθεί το κοινό δυναμικό προγραμματισμού. Θα έλεγα λοιπόν ότι μας ε, ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός, μόλον ότι η δρόμοι που οδηγούν στην πολιτική πάρα πολλές φορές είναι πάρα πολύ πολύπλοκοι και μπορεί να οδηγήσουν σε παράδοξες καταστάσεις. Έχουμε ένα κέντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων το οποίο ε, συνδέεται με μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε ένα προσωρινό κέντρο το οποίο προσπαθούμε να καταστήσουμε μόνιμο κατ' ουσία. Έχουμε ένα ουδέτερο κέντρο από την άποψη του προπολογισμού, αλλά θα πρέπει ε, να έχει πρόσβαση στο προπολογισμό των μη στρατιωτικών ε, δράσεων της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αν θέλουμε να είναι κάτι καινούριο πραγματικά και ουδέτερο από την άποψη του προπολογισμού. Εμείς καταλαβαίνουμε τους λόγους που βρίσκονται στη βάση αυτών των πολιτικών και αυτών των πολύπλοκων διαδρομών. Βεβαίως ευχόμαστε κατ' ουσία να κινηθούμε προς μια πιο αποτελεσματική και σταθερή αύξηση του δυναμικού. Αυτό μας οδηγεί στο να ζητήσουμε ορισμένε διευκρινήσεις, να διατυπώσουμε ορισμένε ερωτήσεις. Από την άποψη την ποσοτική, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικές ενδείξεις, αν βεβαίως υπάρχουν ενδείξεις, αν υπάρχουν προβλέψεις για τον αριθμό των ατόμων, για το επιτελείο, για το προσωπικό, το οποίο έχει περάσει από το ένα επιτελείο στο άλλο, καθώς και τον αριθμό των αποσπασμένων από τις χώρες μέλη. Δεύτερον, αν υπάρχει, αν έχει γίνει κάποια εκτίμηση του κόστους επί του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, βεβαίως, μολον, εμείς είμαστε σαφώς υπέρ του να υποστηρίξει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός αυτή την αυτή την υποδομή. Είμαστε υπέρ του να τα αναλάβει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικά θεωρούμε ότι είναι σωστό. Και βεβαίως ε, τη στιγμή κατά την οποία έχουμε δυνατότητες στα πλαίσια του προπολογισμού για στρατιωτικές ενέργειες, μόνο ότι στην ουσία συνδέεται με μη στρατιωτικές ε, ενέργειες, αναμένουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Δεν ήθελα να καταλάβω καλύτερα τη σχέση με την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, επειδή πρόκειται για μία μη στρατιωτική δράση, η οποία έχει σχέση με αυτό το κέντρο και τη CPCC. Τώρα σε ό,τι αφορά τις δύο επιχειρήσεις, θα ήθελα να γνωρίζω Εάν αυτό το κέντρο επιχειρήσεων θα ήθελε να επιτελέσει και τις δύο αποστολές. Και πώς θα γίνει η κατανομή του προσωπικού. Ποια δεν είναι η σχέση του με την CNPT. Με τον πυρήνα, δηλαδή που ασχολείται με το θέμα του στρατηγικού προγραμματισμού. Ευχαριστώ, κύριο Σέλλερ. Κύριε Στίβενσον, θα ήθελα καταρχάς να σας ε, ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Ε, είδαμε ε, ε, ότι είμαστε ένα χρόνο μετά από τα ψηφίσματα για την συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών ε, δραστηριοτήτων και είχαμε πολύ καλή συνεργασία, έχουμε μια πολύ καλή έκθεση από το, από το Κοινοβούλιο αλλά και από εσάς καλή συνεργασία. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Γνωρίζετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και ένα πρόγραμμα πολιτικής ας πούμε έρευνας και το Κοινοβούλιο κάνει μια συζήτηση για αυτό το πρόγραμμα και υπάρχει και η πρόταση της Κομισιόν για τον ορίζοντα 2020 όπου οι πολιτικές και στρατιωτικές ε, αποστολές είναι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ε, έρευνας. 1,4 ε, ήταν τα δις που τώρα έγιναν 1,7 και έχουμε αυτόν τον προϋπολογισμό 1,7 που θέλουμε να τον φτάσουμε στα 2 δις. Είναι μια νέα αποστολή. Ε, ξέρετε ότι όλα τα προγράμματα έχουν, έχουν συγκεκριμένες αποστολές. Αυτή είναι μια νέα αποστολή και το λέω λίγο προσεκτικά γιατί είμαστε νωρίς στις συζητήσεις. θέλουμε να δώσουμε για αυτήν ε, μισό δις δεν είναι ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα R&D, είναι ένα pre-commercial procurement πρόγραμμα. Διοικητικής μέρημνας δηλαδή, ε, συγγνώμη, προμηθεών. Θα ήθελα λοιπόν ε, να συζητήσουμε μαζί αυτό το θέμα. Γιατί είναι ένα πολιτικό θέμα, το pre-commission procurement, αλλά έχει να κάνει ε, και με τη μισθοδοσία. Ε, από ποιον θα είναι το, αυτό το κομμάτι, από τα κράτη-μέλη, όσον αφορά αυτές ε, τις, οι προμήθειες αυτές, από πού θα προέρχονται, από τα κράτη-μέλη. Άρα, έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς η συνεργασία έχετε με την DG, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας, και μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας θα ήθελα να μάθω περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Σπαλέτσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια υπόθηκε ότι η βασική απειλή για την ασφάλεια είναι οι κλιματικές αλλαγές. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω την εξής ερώτηση. Η κλιματική αλλαγή και οι αναφιόμενες κρίσεις, πότε αυτό θα γίνει πραγματικότητα και σε ποια περιοχή πάνω απ' όλα. Merci, Madame Κόπα. Ευχαριστώ, κυρία Κόπα. Thank you. Thank you, Mr ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση που κάνετε. Η ερώτησή μου δεν με αυτή το προηγούμενο συναδέλφων. Δηλαδή πώς αυτό το επιχειρηματικό κέντρο θα μπορούσε να συνδυαστεί με άλλες αποστολές που αφορούν ε, βοήθεια στην ανάπτυξη, η ανθρωπιστική βοήθεια. Πώς φαντάζεστε αυτή τη συνεργασία, γιατί τότε οι πανίδιοι συνάδελφοι, έχουμε πολύ λιγότερους πόρους και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί σε έναν κόσμο ε, όπου οι προκλήσεις αυξάνονται. Τι, πώς θα συνεργαστείτε με τις μη στρατιωτικές αποστολές. Ευχαριστώ. Κύριε Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό την ανάληψη, την ανάληψη δράσης από το κέντρο. Νομίζω ότι θα είναι σημαντικό και για την Ρουμανία. Έχω μια σύντομη ερώτηση που αφορά τη συνεργασία μεταξύ κέντρου και των άλλων δυνάμεων που αναπτύσσονται στην περιοχή. Το ΝΑΤΟ, οι εθνικέ αποστολέ. Πώ αντιλαμβάνεστε αυτή τη συνεργασία, γιατί είναι απαραίτητο να υπάρξει στενή συνεργασία και να συντονίσουμε τι δράσει μα έτσι ώστε να στεφτούν από επιτυχία οι προσπάθειέ μα. Ευχαριστώ, κύριο Στίβεν, για τι απαντήσει. Και μετά ο κύριο Βανόφσκι, που θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε ορισμένα θέματα. Well, <clears throat> thank you very much. Ευχαριστώ καταρχάς για τις πολύ ενδιαφέρουσες και πολλές ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με μία που θεωρώ ε, πολύ σημαντική. Ε, κάτι που είναι ας πούμε που διανύει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων είναι η βάση της ενεργοποίησης του κέντρου επιχειρήσεων και έχει να κάνει με τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη συνεργασία τους. Εμείς θέλουμε να δώσουμε εμπειρογνωμοσύνη, μακροπρόθεσμα και τώρα έχουμε μια νέα αποστολή, την RNCB, που είναι στην ουσία μη στρατιωτική αποστολή αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτή στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη. Έτσι λοιπόν το κέντρο επιχειρήσεων θα υποστηρίξει στρατιωτικά αυτή τη μη στρατιωτική αποστολή. Στην ουσία θα προσπαθήσει να συνδυάσει τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά στοιχεία. Και τώρα υπάρχει μια τεχνική αποστολή στην οποία θα πάω, γιατί έχουμε στο Συμβούλιο, από το Συμβούλιο λάβει την έγκριση. Ε, έχουμε μια τέτοια αποστολή λοιπόν που συνδυάζει αυτή τη στρατιωτική και μη στρατιωτική ε, διάσταση και έχουμε ε, στο τέλος ε, του μήνα ε, κάτι που περιλαμβάνει και στρατιωτικούς και με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό σημαίνει επίσης ότι υπάρχει ένα σύνδεσμος με την Κομισιόν. Ο Μαρτιν Σούμπεν είναι αυτός που ήταν πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι εκεί στο πίσω μέρος της αίθουσας και ήρθε στην ε, περιφέρεια για να γίνει μια διάσκεψη με τους ανθρώπους εκεί ε, και να πω για την Κομισιόν ότι υποστηρίζουν πολύ το πρόγραμμα μας ε, και τώρα το ΜΑΣ και η RNCP αποστολή θα συνδυαστούν έτσι ώστε το ΜΑΣ να μπορέσει να χρηματοδοτήσει εξοπλισμό, κάποια ε, μαθήματα εκπαίδευσης κτλ. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν φροντίζει για τη σταθερότητα. Ήταν ε, μια κατευθυντήρια γραμμή, αλλά και ε, πέρα από τα σύνορα. Γιατί το ΝΑΤΟ, ας πούμε, συνεργάζεται όταν μιλάμε για δημιουργία υποδομής, τα Ηνωμένα Έθνη, UNDP, και άλλοι οργανισμοί που ας πούμε εκπαιδεύουν αστυνομικούς ε, ή ε, άλλες ε, μονάδες έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η αποστολή. Στην ουσία συγκολούμε διάφορα διεθνή εργαλεία και ευρωπαϊκά εργαλεία έτσι ώστε να αυξηθούν τα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο έργο, ένα πρόγραμμα ε, το οποίο στηρίζεται από το επιχειρησιακό ε, κέντρο, ε, το οποίο είναι αυτό που συνδυάζει τους εμπειρογνώμονες, τους συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τους εμπειρογνώμονες από όλους τους τομείς. Επίσης, έχουμε και ένα σχέδιο ε, δράσεις. Έχουμε το κέρας της Αφρικής, μια στρατηγική εκεί ευρεία και διάφορες αποστολές. Θέλουμε όμως έναν σύνδεσμο, ε, ο οποίος ε, θα κάνει όλα αυτά τα στοιχεία ένα σχέδιο δράσης. Μια εκστρατεία, όπως τη λέμε. Έχουμε λοιπόν σε επίπεδο επι, επιτελεί ολοκληρώσει ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Θα πάμε ένα επίπεδο παραπάνω και θα ξεκινήσουμε τις διαβουλεύσεις της υπηρεσίας για να γίνει πιο επίσημο και να συνδυαστούν όλα αυτά στα στοιχεία. Η όλη προσέγγιση στο κέρας της Αφρικής είναι στην ουσία μία εικόνα για το τι μπορεί να συμβεί, μια δοκιμαστική περίπτωση ε, που μας βοηθά ε, να δούμε τι θα γίνει όταν μια ολοκληρημένη προσέγγιση πραγματοποιείται. Θέλουμε λοιπόν ε, να δούμε τι θα γίνει ε, ε, όταν λειτουργήσει το όλο πράγμα που είναι πιο δύσκολο και καθημερινό. Αυτά για τη στρατιωτική και μη στρατιωτική συνεργασία που είναι ε, στο κέντρο αυτής της επιχείρησης. Για την ερώτηση του κύριου Έλερ, δεν γνωρίζω 100% τα... το πρόγραμμα αυτό της μη στρατιωτικής ασφάλειας. Μας έχουν κάποια στιγμή προσκαλέσει. Ε, επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την συνεργασία μέσα στα πλαίσια της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Ε, επίσης, μέσα στα μετά από μια πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης ε, Βιομηχανίας ε, ε, θα συναντηθούμε και μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας θα συνεργαστούμε ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργαστούν. Συγγνώμη που διακόπτω, δεν έχει να κάνει με τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Τώρα γράφουμε μια νέα αποστολή για το πρόγραμμα. Είναι η συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Θα γίνει έρευνα ε, σε στρατιωτικό επίπεδο. Ε, δεν είναι μάλλον σε στρατιωτικό επίπεδο η έρευνα, γιατί δεν υπάρχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο γι' αυτό, αλλά για μη στρατιωτικέ αποστολέ, αν έχουμε λοιπόν ένα επιχειρησιακό στρατηγείο, για αυτά θα μπορούμε να ξοδέψουμε ε, τα χρήματα για το R&D και για το pre-commercial procurement. Αυτή είναι η ιδέα. Δεν έχει να κάνει με τον οργανισμό. Και ρωτάω τώρα, εφόσον φτάνουμε σε, αυτή τη, σε αυτό το στάδιο της πιο ενισχυμένης συνεργασίας, να πω ότι ε, δεν πάει μέσω του οργανισμού. Χρειάζεται άμεση εμπλοκή από εσάς. Ναι, ευχαριστώ. Θα προτείνω στο επιτελείο μου να εργαστούμε λίγο παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν γνωρίζω επαρκώς όσα λέτε. Ε, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει το CSTP να εμπλακεί, δηλαδή η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Συμφωνώ με την κυρία Νικολάη, ε, η Αταλάντα και όσοι συνεργάζονται με την Αμερικανική ε, πλευρά. Ε, τα στρατηγία των δύο επίσης ε, συνεργάζονται και υπάρχει και ένας ε, Ολλανδός συνάδελφος από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Η παρουσία του ΝΑΤΟ είναι περιορισμένη αυτή τη στιγμή. Μόνο ένα πλοίο ή δύο έχουν μείνει. Έχουν όμως σημαντική συμβολή σε επίπεδο τεχνολογίας. Αλλά για άλλη μια φορά η ενεργοποίηση του κέντρου επιχειρήσεων θα πρέπει ε, ε, να έχει να κάνει όχι μόνο με την Αταλάντα και το αλλά και με τις τα άλλα σημεία, τα άλλα στοιχεία της ε, όλης προσέγγισης. Μετά έχω πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, σχετικά με κάποια νούμερα. οι άνθρωποι θα εργάζονται σε αυτό το επιχειρησιακό κέντρο. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πω. Θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των υπευθύνων, αυτή τη στιγμή έχουμε το EUTM, το οποίο ε, ήδη ε, έχει δύο άτομα, την ομάδα σύνδεσης για την Αταλάντα, δύο ή τρία άτομα, συνολικά πέντε λοιπόν. Και άκουσα ότι σε μια αρχική φάση αυτοί που θα πάνε στην τεχνική αποστολή για την ε, προετοιμασία του RMCB θα είναι 6 με 7 εμπειρογνώμονες. Είναι η φάση σχεδιασμού και μετά έχουμε τη φάση διεξαγωγής γιατί θα γίνουν σε δύο φάσεις οι επιχειρήσεις, άρα αν τους μετρήσουμε θα φτάσουμε σε ένα νούμερο 10-15 άτομα. Αλλά αυτό είναι κάτι που αδρά εγώ έτσι και ε, πολύ πρόχειρα υπολογίζω. <coughs> Δεν έχω επίσημες πληροφορίες. Σε επίπεδο κόστους, το αρχικό κόστος θα είναι πολύ λίγο νομίζω. Γιατί την εμπειρογνωμοσύνη τη δίνει το στρατιωτικό επιτελείο. Αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποια στοιχεία σε αυτό το επίπεδο που δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, τα κράτη-μέλη θα δώσουν ε, από την πλευρά τους τα χρήματα. Ε, τώρα, ποιες είναι οι σχέσεις με την CPCC εφόσον αυτή η δημιουργία ναυτικών δυνατοτήτων είναι ε, ένα μη στρατιωτικό ε, θέμα, έχουμε τον ε, διοικητή και το επιχειρησιακό κέντρο θα υποστηρίζει το στρατιωτικό κομμάτι της εμπειρογνωμοσύνης και θα υπάρχει αυτή η συνέργεια ιδανικά και θα έρθω σε αυτό το ερώτημα. Φυσικά Έχουμε και τα ε, μη στρατιωτικά στοιχεία της αποστολής RMCP εκεί. Ο ένας κάθεται στην αριστερή πλευρά του διαδρόμου, ο άλλος στη δεξιά. Χρησιμοποιούν ε, τις ίδιες αίθουσες συνεδριάσεων. Συνεδριάζουν κάθε μέρα. Υπάρχει, ας πούμε, μια συγκατοίκηση που δημιουργείται συνέργειες. Άρα η σχέση είναι πολύ στενή. Φυσικά το επιχειρησιακό ε, κέντρο βρίσκεται εκεί και για τις άλλες δύο στρατιωτικές αποστολές. Και φυσικά θα θέλαμε να δούμε μια πιο έναν πιο ευρύ σχεδιασμό, μια πιο ευρία αρχή σχεδιασμού στρατιωτικών με στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά νομίζω ότι αυτό το κέντρο είναι ούτως ή άλλως κάτι σημαντικό, μια καινοτομία. αλλά αυτό το κέντρο σχεδιασμού θα ασχολείται όχι μόνο με το κέρας της Αφρικής και με άλλες περιοχές. Είναι όμως σημαντικό που έχει έναν σημαντικό στόχο, όχι μόνο την υποστήριξη, αλλά και τη δημιουργία συνεργειών και τη συνεργασία. Η διάρκεια είναι ακόμα υποδιαπραγμάτευση, συζητείται. Ξέρω ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν τη δική του συλλογική το καθένα τέλος πάντων, κοινοβουλευτική και μη ε, κοινοβουλευτική, λεκτική και μη. Συνεχίζεται η συζήτηση και γι' αυτό δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Έχουμε προτείνει κείμενα που φαίνεται ότι λειτουργούν και άλλα όχι. Όλοι συμφωνούν ότι επί της αρχής έχει ενεργοποιηθεί για όλη τη διάρκεια. Χρειάζεται μία αναθεώρηση ε, να δούμε αν τα πράγματα, μια επισκόπηση ενδιάμεση για να δούμε αν τα πράγματα πάνε καλά και ούτω καθεξής. Να πω και κάτι άλλο. Πότε μπορούμε να κλείσουμε τον όρο και να περάσουμε τα, αυτά στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή όχι. Όχι. Μάλιστα. No, this is not the case yet. No, no, not yet. Κοιτάξτε, η λογική είναι ότι δημιουργήθηκε και να υποστηρίξει τις αποστολές της LCB. Και βεβαίω το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρξει μια διασύνδεση με τις άλλες στρατιωτικές αποστολές. Ήδη έχουμε ένα επιχειρησιακό κέντρο για τις αποστολές στην Αταλάντα. Βεβαίως, για να μεταφερθεί στις Βρυξέλλες χρειάζεται πολιτική συμφωνία και δεύτερον, νομίζω ότι θα, χρειαστεί, θα χρειαστούν πολύ περισσότερα χρήματα. Νομίζω ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα για να ενεργοποιηθεί αυτό. Υπάρχουν ε, κομπιούτες, υπάρχουν τραπέζια, υπάρχουν καρέκλες, υπάρχουν οι άνθρωποι. Τώρα το θέμα είναι να δραστηριοποιηθεί. Ενδεχομένως ε, μιλάμε για αυτό που βλεπόταν από την αρχή βρίσκεται εκεί για να υποστηρίξει την αποστολή και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί έχει αλλάξει το όλο πνεύμα. Υπάρχει αυτή η ενοποιημένη, η γενικότερη προσέγγιση και πιστεύω ότι αυτό το κέντρο επιχειρήσεων μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένω μακρηγόρησα, ενδεχομένω ξέχασα να απαντήσω σε ένα-δύο ερωτήματα. Ε, αναφέρθηκε ένα αρκετά δύσκολο ε, θέμα. Νομίζω ότι οι χώρες μέλη θα επιδείξουν την ίδια διάθεση συνεργασίας στην ανέβρεση λύσεων. Βεβαίως μέσα στα υπάρχοντα πλαίσια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στρατηγός. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιστρέφω Τώρα το επιτελείο ε, βρίσκεται στα πλαίσια της, ε, των υπηρεσιών εξωτερικής δράσης. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να πω δύο λόγια για το επιχει... κέντρο επιχειρήσεων. Εγώ μετά τον κύριο Στίβενς θα ήθελα να πω εν συντομία ότι πιστεύω ότι τι είναι το ότι βρέθηκε ένα συμβιβασμό μεταξύ των διαφόρων απόψεων και η κοινή βάση είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τον συντονισμό, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί για να βασιστούμε σε κοινέ δομέ. Αυτό ακριβώ θα κάνουμε τώρα. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα. Θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το συμβιβασμό και να τον καταστήσουμε λειτουργικό. Και τρεις ε, βασιτές, βασικές αρχές ε, που προήλθαν από τις χώρες μέλη εμπεριέχονται σε αυτή την ε, απόφαση. Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Βόλτ Στίβενς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που μου ζήτησε να αναπτύξω ο πρόεδρος της δραστηριότητας του ΙΟΜΕΣ, την τελευταία φορά που επισκέφθηκα την Επιτροπή πρόβλεψα ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν με τρόπο θετικό. Συνεχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει μία θετική τάση ακόμα. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι εύκολα γιατί έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές προσεγγίσεις, με διαφορετικό τρόπο εργασίας, αλλά πιστεύω ότι γινόμαστε καλύτεροι βδομάδα με τη βδομάδα. Το μήνυμα μου απευθύνεται και προς το στρατιωτικό σκέλος, προς στρατηγικού ε, που συναντάω και που συχνά απευθύνουν ερωτήσεις κατά πόσον αυτό είναι λειτουργικό. Ναι, είναι λειτουργικό. Η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκυται στο ότι μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί πιο ουσιαστική γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που συντονίζονται από τον πρέσβη κ. Στίβενς στα πλαίσια του ESDP αλλά και οι νέες διαδικασίες ε, που έχουν σχέση με τον ειδικό εντεταλμένο προσώπου, προσώπους όλων των φορέων που θα μπορούσαν να, να έχουν κάποια σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Σε όλη μου τη ζωή εργάστηκα σε διάφορες οργανώσεις και στο ΝΑΤΟ και σε μη στρατιωτικέ οργανώσεις. Πάντοτε μιλάμε για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Για πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει από την αρχή και καταλήγουμε σε καλύτερες αποφάσεις σαν αποτέλεσμα αυτού. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, δεν θα ήθελα να πω το τι συνέβη πέρσι. Αυτό όμως είναι αλήθεια. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του Πακιστάν, της ε, Λιβύης, ε, του κέρατος της ε, Αφρικής. Όλα αυτά αποτελούν πολύ καλά παραδείγματα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Βοσνία Ερσεγοβίνη, όπου όχι μόνο οι στρατιωτικοί έχουν ένα μέσον, αλλά και η Επιτροπή και διάφοροι επίτροποι δραστηριοποιούν ποιήθηκαν και υπήρξε ε, συντονισμός και στις Βρυξέλλες και επί τόπου. Αυτό, αυτά όλα μας έχουν καταστήσει περισσότερο ουσιαστικούς, περισσότερο αποτελεσματικούς, δίχως να υπάρξει μια παράλληλη αύξηση του κόστους. Το κόστος παραμένει το ίδιο, η αποτελεσματικότητα όμως αυξάνεται. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να παραθέσω παραδείγματα. Εγώ σας παρέθεσα μερικά, βεβαίως ε, η σειρά σας να κάνετε ερωτήσεις αν θέλετε. Μετά θα έχω την ε, δυνατότητα να σας εξηγήσω πώς εφαρμόζονται όλα αυτά και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται περισσότερο αποτελεσματική. Αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι ενδιαφέρον ε, είναι το θέμα του συντονισμού σε διάφορα επίπεδα. Βλέπω ότι στα πλαίσια αυτού του συντονισμού ε, χώρες που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν προσπαθούν να οργανώσουν συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Ε, μια προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των μεμονωμένων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρξει δηλαδή ένα συντονισμό σε στρατιωτικό επίπεδο πάλι, ένας ευρύτερο συντονισμό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επίσης έχουν αλλάξει την ε, στάση τους έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας ε, συντονισμό σε στρατιωτικό επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει με την Κίνα και τη Ρωσία που τους ενδιαφέρει ε, ιδιαίτερα το θέμα της συνεργασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό μου ρόλο, ο Γενικός Διευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου έχω δύο ρόλους και το δύο ισχύει και στον ΝΑΤΟ. Το βλέπω το θέμα από την προοπτική των επικεφαλής άμυνας, το βλέπω από την άποψη των μελλοντικών δυνατοτήτων και των επιχειρηματικών αναγκών. Εκεί εστιάζω την προσοχή μου. Εγώ όμω αναφέρομαι στον ύπατο εκπρόσωπο, στην ύπατη εκπρόσωπο, στην ουσία καταλήγω σε ορισμένα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στο πρέσβη Στίβεν. ή στον υπεύθυνο τη γεωγραφική περιοχή που αναπτύσσει μια στρατηγική πλαίσιο για μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Μόνον αν αυτά τα έγγραφα γίνουν δεκτά από την ύπατη εκπρόσωπο, περνάνε στην πίση και μετά γνωμοδοτεί η Στρατιωτική Επιτροπή. Μερικές φορές ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Για μένα είναι πολύ πιο εύκολο το να γράψω ένα έγγραφο. Αν θέλετε, ω στρατιωτική να έχετε μια γενικότερη προσέγγιση, θα πρέπει να δεχτείτε ότι θα πρέπει να γράφετε έγγραφα που είναι ολοκληρωμένα. Έτσι ώστε να μπορούν να έχουν άποψη όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι καλύτερα και πιο σοφά βέβαια, πιο συνετά παρέθεσα παραδείγματα σε ό,τι αφορά τις διάφορες επιχειρήσεις. Ο άλλος μου ρόλος, το να υποστηρίζω και να βλέπω ε, το θέμα ως επικεφαλής της άμυνας, αυτό το κάνω σε στενή συνεργασία με τον πρέσβη Walter Stevens, που είναι υπεύθυνο για θέματα συνεργειών. Ένα από τα θέματα που ετέθησαν από μερικούς από εσά. Επίσης, έχω πολύ καλή συνεργασία με την EDA, όπου ε, παρέχω τις στρατιωτικές μου ε, γνώσεις και εκεί υπάρχει καλό συντονισμός με το ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε επίπεδο ICT. Είναι ενδιαφέρον να καταλάβουμε τη διαφορά. Ποιος κάνει τι. Η ICT το ΝΑΤΟ, το Νόρφογκ είναι υπεύθυνα και για τον εντοπισμό όλων των επιχειρησιακών απαιτήσεων, κάτι που μεταφράζεται σε προγράμματα, εγώ περιορίζομαι στο ρόλο του επικεφαλής της άμυνας. συγκεντρώνω τα όσα έχουμε μάθει από τις επιχειρήσεις. Τα συζητάμε και προσπαθούμε να υπάρξει μια κοινή άποψη για την οποία θα ενημερώσουμε την EDA. Η EDA είναι εκείνη η οποία δίνει κάποια συνέχεια σε αυτό το project, σε αυτό το έργο. Παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά. Στην ουσία εμείς αναζητάμε συνέργειες, υπάρχουν αρκετά προγράμματα ε, τα οποία έχουν πάντοτε κάποιον επικεφαλής. Ένα άλλος, ένας άλλος τομέας είναι το pooling and sharing. Ε, κοινές, ε, κοινή πόρη και καταμερισμός αυτών των πόρων. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα την ανάλυση που γίνεται εδώ αυτό που δεν είναι σαφές είναι αυτό που το επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει σε ό,τι αφορά το σημείο αυτό. Δηλαδή το ΤΣΟΤ μέσω της Στρατιωτικής Επιτροπής λαμβάνει πρωτοβουλίες. Εμείς προσπαθούμε να εναρμονίσουμε όλα αυτά. Να σας παραθέσω ένα παράδειγμα. Στην πρώτη φάση, πέρσι, όταν ε, έγινε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τα καλά, προγράμματα για pooling and sharing, δεχτήκαμε 300 πρωτοβουλίες. Τα αναλύσαμε, αναλύσαμε πέντε κριτήρια. Ένα βεβαίως αφορούσε την εξοικονόμηση κόστους, το θέμα ε, των ε, προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα των υποδομών και των δυνατοτήτων, εάν ε, γίνουν σεβαστά όλα τα κριτήρια, τότε το project θα στραφεί από επιτυχία. Υπάρχουν χώρες μπέλη που ήθελαν να έχουν τις υποδομές, αλλά που δεν ήθελαν να ασχοληθούν ε, οι ίδιες. Όλα αυτά είναι παραδείγματα. Αν υπάρχουν πιέσεις καταλαβαίνουμε ότι εάν θέλουμε ε, να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας θα πρέπει να συνεργαστούμε. Υπάρχουν τρεις άλλες χώρες που θέλουν να ενταχθούν και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια χώρα που είναι επικεφαλής. Πιστεύω ότι πολλές χώρες πληρούν ε, τα κριτήρια, αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί μια τέτοια χώρα και ασκούμε πιέσει στι διάφορε χώρες για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό για τα διάφορα προγράμματα. Ένας άλλος τομέας που δεν συνδέεται πάντοτε με το EDA αφορά το τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Υπάρχουν δύο είδη πρωτοβουλίων, πρωτοβουλίες, τις οποίες διαπιστώνουμε ότι χρειαζόμαστε κοινέ υποδομές, ε, κοινέ ε, δαπάνες, κοινή τεχνολογία. Όλα αυτά γίνονται προγράμματα και τα υποβάλλουμε στο EDA. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι το να εντοπίζουμε και σήμερα το απόγευμα στη Στρατιωτική Επιτροπή θα συζητήσουμε αυτές ε, τις λεπτομέρειες, δεν θα επισέλθω λοιπόν τώρα σε αυτά τα σέματα. είναι δυνατόν δίχως τεχνολογική ανάπτυξη, χωρίς συγκεκριμένα προγράμματα, να βρούμε το μίσο που μπορούμε να συνεργαστούμε και να εξοικονομήσουμε. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτού σε πολλές χώρες η χρήση των αεροσκαφών μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε η χρήση των ελικοπτέρων. Έρχεται μια στιγμή που σταματάει κανείς να λειτουργεί μια σχολή, γιατί υπάρχουν άλλοι που έχουν τις υποδομές και το επιβεβλημένο είναι συνεργασία. Αυτό μπορεί να το κάνει κανείς και σε άλλους τομείς. Αυτός είναι ένας τομέας όπου το στρατιωτικό επιτελείο θα μπορούσε να βρει με μεγαλύτερη ευκολία χρήματα σε αντιπαράθεση με τα συγκεκριμένα project που απαιτούν πολλά χρήματα. Δύο λόγια για το θέμα της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είμαι ευγνώμων που μπορούμε να έχουμε ένα συντονισμό, έναν άτυπο συντονισμό μεταξύ επιτελείων με το ΝΑΤΟ θα ήθελα να σας πω όμως ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Μπορούμε να ενημερώσουμε η μεν τους δε ποιος κάνει τι και μετά ε, συζητάμε ποιος μπορεί να κάνει το κάθε τι καλύτερα δεν λέω ότι δεν υπάρχει καμία επικάλυψη γιατί ορισμένες χώρες μέλη θέλουν να προωθήσουν τα προγραμματά τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ατλαντική Συμμαχία. Αλλά δεν υπάρχει επικάλυψη. αυτό θα παραμείνει μια επιλογή των χωρών μελών. Αυτό που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό στην όλη συζήτηση που γίνεται για το pooling and sharing, διευκολύνουμε τις χώρες μέλη και δημιουργούμε όσο γίνεται περισσότερες ε, υποδομές για τις χώρες μέλη. Δεν μιλάμε για υποδομές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των μεμονωμένων χωρών Και οι χώρες μέλη αποφασίζουν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν, είτε σε εθνική βάση, είτε σε βάση ε, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Συνεπώς και συμφωνώ με την έκθεσή σας όταν αναφέρεστε στο Ευρωπαϊκό Επιτελείο Μεταφορών. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πολλές χώρες συνεργάζονται, αυξάνουν το κοινό τους δυναμικό, τις κοινέ τους υποδομές, αλλά οι χώρες μέλη αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις υποδομές. Είτε αυτό θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε εθνική βάση, σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ κτλ. Το ίδιο Ισχύει και με την, ε, το αεροπορικό επιτελείο στην ε, Ουγγαρία. Οι χώρες μέλη αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιηθεί το κάθε τι. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχουν δυσκολίες ό,τι αφορά το θέμα του pooling and sharing. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία ακόμα, γιατί πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της συζήτησης άκουσα για την δυσκολία που αντιμετωπίζουν ε, τα μέλη που λένε ότι ναι, αλλά θα χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι η κυριαρχία συνεπάγεται την ελευθερία στην απόφαση και την ικανότητα στη δράση. Γιατί δεν έχει νόημα να μπορεί κανείς να αποφασίσει να κάνει κάτι, αλλά να μην μπορεί να το κάνει. Τότε δεν έχει κυριαρχία και αν ο μοναδικός τρόπος για να αποκτήσει κανείς τις υποδομές για να δράσει είναι μέσω της συνεργασίας με τους άλλους, τότε δεν παραχωρεί κανείς κυριαρχία, αλλά κερδίζει κυριαρχία. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου δουλειά. Κατόπιν αιτήματος του Τσότ, πώς θα βρούμε τις πρωτοβουλίες όπου είναι χρήσιμη η συνεργασία και αν φτάσουμε σε ένα project να το δώσουμε στην EDA και να μπορέσουμε να βρούμε, να επιτύχουμε συνέργειες στα πλαίσια της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Εκεί δεν χρειαζόμαστε ένα project και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε επίσης να κάνουμε σταματήσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σα για οποιαδήποτε ερώτηση. Euh, κύριε πρόεδρε, ε, κύριε Τσάτικε μου θα είχα μια ερώτηση, λέει ο Πρόεδρο, σε ένα σημείο πάρα πολύ πρακτικό. Για να έρθω στο τη Αφρική, αυτή η Αταλάντη, η Αταλάντα, είναι πολύ εμβληματική για την ΕΕ σε στρατιωτικό επίπεδο, στρατηγία μου εκτός από τις πολιτικές δυσκολίες που γνωρίζουμε όσον αφορά την νομική διαχείριση της πειρατείας, της πειρατείας από τις κατευθύνσεις Σομαλία. Ωστόσο παραμένει ένα θέμα το οποίο παραμένει σαν πρόβλημα για εμάς τους δηλαδή πώς είναι ικανή η Ευρώπη να διαθέτει εκεί δυνάμεις διότι οι χώρες είναι όλο και περισσότερες επιφυλακτικές για την κινητοποίηση και στην επιστράτευση ανδρών οι οποίοι θα ήθελαν εκεί πέρα να επανδρώσουν αυτές τις δυνάμεις. Νομίζω πως είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία συζητείτε και βεβαίως είναι μία από τις αποστολές τις πιο εμβληματικές της ΕΕ. Πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες μας και Ε, και βεβαίω θα θέλαμε την άποψή σα τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε, τι λείπει, τι είναι λοιπέ, τι δεν είναι σωστό. Είναι πάρα πολύ ε, η εξειδικευμένη αυτή η ερώτηση που σα κάνω. Ο κ. θα ήθελα να παρέμβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, στρατηγία μου. Πώς να το καταθέσω τώρα αυτό. Για να κάνουμε τις δραστηριότητες μας πολύ πιο αποτελεσματικές, έχουμε προβλέψει έχουν προβλέψει την μεταρρύθμιση του προγράμματος Αθηνά. Υπήρξαν ε, αποτελέσματα. Πώς εσείς λοιπόν βλέπετε την παρούσα κατάσταση. Αυτές οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι σωστές. Καθώς επίσης η δυνατότητα μεταφορών είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση. Είστε ικανοποιημένο από τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερη ερώτηση ως αυτό το pool and sharing, συγκεντρώνω και διαμοιράζω. Μιλήσατε λοιπόν για πέντε κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται προκειμένου. Υπάρχει επί, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αυτό το πράγμα και κατά πόσο διαρωτώ με εσείς είστε διατεθειμένος ή εκπλήσεστε ότι ορισμένα πράγματα κατατίθενται σαν project και μήπως θα, θα μπορούσαν να μπορούν, να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα στα πλαίσια της ΕΕ και αν αυτό συμβαίνει πραγματικά ποια θα, ποιο θα ήταν το κίνητρο σας, διότι το βασικό θέμα είναι να προχωρήσουν τα πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οι παρατηρήσεις που κάνατε είναι ενδιαφέρουσες πρωτίστως, γιατί όπως γνωρίζετε καλά, αυτή η υποεπιτροπή ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την έννοια του compressive approach. Εμείς είμαστε σαφώς θειασότες αυτής της άποψης και Βλέπουμε με χαρά το γεγονός ότι κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση μεταξύ των άλλων επιλογές για τις οποίες, τις οποίες εμείς είχαμε στηρίξει. Αναφέρουμε το θέμα του μηχανισμού συνεργασίας πολλών φορέων. Μας περιγράψατε μία ένα μηχανισμό λειτουργικού χαρακτήρα, μια δυναμική θεσμική που θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας πολιτικής. Βεβαίως, στα πλαίσια της ασφάλειας και της άμυνας, μας ενδιαφέρει να διαπιστώσουμε αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε κινητοποιήσει λειτουργικές και διοικητικές ε, διοικητικούς μηχανισμούς. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε από πλευρά χωρών μελών να συνεχίζει να παρατηρείται μία άρνηση ε, υιοθέτηση αυτού του δρόμου. Στην ουσία είναι τι θα επικρατήσει στο τέλος, αν αυτή η δυναμική είναι επαρκής για να αντισταθμίσει μια έλλειψη πολιτικής βούλησης που σήμερα είναι σαφής, αντικατοπτρίζεται και στα προβλήματα που αναφέρθηκαν και που αφορούν τις διάφορες δυνάμεις. Θα ήθελα να κάνω και μερικές συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πώς λειτουργεί αυτό το αποκαλούμενο crisis platform θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το ρόλο των δομών CSPD. Και αυτό σε σχέση με τις συγκεκριμένες κρίσεις ε, που ε, παραθέσατε. Δηλαδή, πώς ακριβώς ε, αναπτύσσεται αυτή η σχέση μεταξύ των δομών διαχείρισης κρίσης της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και των άλλων ε, ε, τρόπων αντιμετώπισης αυτής της crisis platform, της crisis management board, σε εβδομαδιαία βάση. Στην ουσία μιλάμε για τις ίδιες πλευρές του ίδιου και σε ό,τι αφορά το situation room ε, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ε, ε, ενίσχυση αυτής της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων. Τέλος, ε, με ενδιέφερε ιδιαίτερα αυτό που αναφέρεται, το μιλ του μιλ, η συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών τομέων, μιλώντας για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Αναφερθεί στραφτήκατε σε μια καινούργια στρατηγική εκπροσώπηση στην Ευρώπη χωρών που θα επιθυμούσαν να έχουν μια σχέση μαζί σας. Ε, ποιες είναι οι χώρες που έκαναν αυτή την επιλογή, αυτή είναι η ερώτηση. Merci, Ευχαριστώ. Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ξέρουμε όλοι μας ότι πόσο σημαντική είναι αυτή η εθνικιστική αντιμετώπιση της στρατιωτικής πολιτικής. Δυστυχώς, ξέρετε, γίνεται όλο και πιο σημαντική στο διάλογο τον οποίων έχουμε όλων. και αυτή τη στιγμή θέλουμε να έχουμε περισσότερη βάρος στο τοπικό επίπεδο και βεβαίως εσείς έχετε δύναμη αυτή τη στιγμή να ισορροπήσετε τα πράγματα και να έχετε μια κοινή προσέγγιση προς τα θέματα. η ερωτήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την ποιότητα του προσωπικού του επιτελείου καθότι για να επιτύχουμε τους στόχους μας ξέρετε ότι υπάρχει το multiculti το πολιτισμικό. Το προσωπικό σας πώς το προσλαμβάνετε είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι σχέση με την πληροφόρηση που πρέπει να υπάρχει γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς οργάνωτε, πώς αυτή ο τομέας πληροφόρησης διοργανώνεται, οργανώνεται, στοιχειοθετείται και επίσης επί του πεδίου αυτοί οι οποίοι είναι οι μάχημοι. Πώς ακριβώς αυτοί οι μάχημοι διαρθρώνονται, πώς αντιδρούν σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Στρατηγέ μου, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Το κέρας της Αφρικής ε, και η συγκεκριμένη ερώτηση για την Αταλάντα δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής ε, βούλησης, αλλά και γεγονός ε, της ζωής ότι όλοι έχουμε οικονομικά προβλήματα και έχουμε και ένα μικρότερο προϋπολογισμό στο επίπεδο της άμυνας και πρέπει να δούμε πώς θα βελτιστοποιήσουμε τη χρήση του. Θα έχουμε λίγα δύσκολα χρόνια μπροστά μας, ελπίζω να είναι λίγα για να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της ασφάλειας και της άμυνας, είναι όλων των τομέων διακυβέρνησης. Είναι ειδικά πρόβλημα λοιπόν των χωρών. Και αν ρωτήσετε εμάς και τον διοικητή, ε, φυσικά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα πράγματα. Η Αταλάντα έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ε, αυτό βέβαια δεν, δεν είναι σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Η μεγαλύτερη λοιπόν προτεραιότητά μας και πρώτη προτεραιότητά μας έχει καλυφθεί. Επίσης έχουμε ε, συμβάλλει στην ασφάλεια και την, ε, σε όλη την περιοχή. Είναι μεγάλη προτεραιότητα για τον Αμαζόνιο ε, γιατί υποστηρίζεται μέσω του EUTM και μέσω από το TFG στο Μογκαντήσου. Έτσι λοιπόν με την υποστήριξη στο Amazon έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη της ασφάλειας εντός της Σομαλίας. Μπόρεσε και αυτό να το καλύψει λοιπόν. Κάποιες φορές ε, πρέπει να θέσει αρνητικές προτεραιότητες ε, σε σχέση με τη συμβολή όλων των άλλων εταίρων. Έχουμε έναν ε, κοινό μηχανισμό με το ΝΑΤΟ και την Συμμαχία των προθήμων της Ευρω... της... Ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ε, παρόλο λοιπόν που προσπαθούμε όσο μπορούμε υπάρχουν πειρατικές δράσεις εναντίον εμπορικών πλοίων την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια τέτοια περίπτωση με ένα πλοίο που θεωρείται ότι ήταν σε έρημνα, ήταν στρατιωτικό τελικά, συνελήφθησαν όλοι. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά έχει τη δυνατότητα να κάνει όλο και περισσότερες τέτοιες ε, δράσεις. Αλλά η στατιστική δείχνει ότι έχουμε λιγότερη επιτυχία από ό,τι είχαμε πέρυσι. Έχουμε αυξανόμενο αριθμό ε, προβλημάτων, ε, μάλλον η πειρατεία έχει αυξηθεί, όμως ε, αν συγκρίνουμε με πέρυσι, έχουμε 25% διαφορά σε σχέση με το 2010. Και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί θα είναι δύσκολο ε, και στο υπόλοιπο έτος να έχουμε όλες τις ε, ικανότητες και υποδομές που θέλουμε. Έτσι λοιπόν άλλαξε τακτική και χαίρομαι τώρα που έχουμε την ε, συμφωνία του να χρησιμοποιηστεί σωματική προστασία και με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή οι χώρες που το θέλουν μπορούν με την εντολή του να, έχουμε, να έχουν αυτή την προστασία σε, στο ίδιο το πλοίο, όχι μόνο ε, συνοδεία από φρεγάτα. Έτσι η φρεγάτα μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ελευθερώνεται. Επίσης, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την ιδιαίτερα δαπανηρή ναυτική επιχείρηση και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε όλες αυτές τις ε, ε, δράσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η δημιουργία δυνατοτήτων ε, σε ναυτικό επίπεδο είναι μία από αυτές, η δημιουργία του επιχειρησιακού κέντρου και η δημιουργία ακτοφυλακής και αστυνομίας εναντίον των ε, ε, εγκληματικών πειρατικών δράσεων ε, στις ίδιες τις χώρες, οι οποίες θα πρέπει στο τέλος να φροντίζουν μόνες τους το πρόβλημα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο και είναι ένας άλλος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συνεχίσει η Αταλάντα. Ο μηχανισμός Αθήνα. Αθήνα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ε, πρωτοβουλία για να υπάρξει βελτίωση εκεί. Όμως η μόνη βελτίωση που υπήρξε είναι αυτή η συμφωνία ο, ο, διαχειριστής να μπορεί να έχει συμφωνίες πλαίσιο όπως ονομάζεται από ό,τι θυμάμαι με εμπορικές και άλλες οργανώσεις που μπορούν να δώσουν υποστήριξη. Γινόμαστε λοιπόν πιο αποτελεσματικοί. Αυτό είναι ένα όφελος. Ελπίζω προσωπικά ότι θα υπάρχουν βελτιώσεις και στην κοινή χρηματοδότηση. Νομίζω και μπορώ να σας πω από την εμπειρία ότι θα ακούσατε ε, πολλές, ε, πολλά επιχειρήματα ότι η ομάδα Β δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Όμως πάντοτε, αν ε, δούμε τα επιχειρήματα, αυτά σχετίζονται σχεδόν πάντοτε με το οικονομικό. Αν κανείς λοιπόν παραπονείται ότι δεν χρησιμοποίησαμε τις ομάδες Β. Την ίδια στιγμή το ίδιο άτομο είναι κατά της κοινή χρηματοδότησης, τουλάχιστον της στρατηγικής ανάπτυξης και επανανάπτυξης της ομάδας. Οπότε πάντοτε έχουμε κάποια κράτη-μέλη τα οποία είναι ενεργά στην ομάδα και κάποιες φορές δεν έχουν καν επιλογή να πούν όχι. Γιατί ο προϋπολογισμός τους δεν μπορεί να ταιριάξει με το υψηλό κόστος όταν πρέπει η ομάδα να πάει σε μεγάλες αποστάσεις για παράδειγμα. Το στρατηγικό κόστος είναι μεγάλο. Και αν πρέπει κάτι να μπει στο προϋπολογισμό θεωρώ ότι δεν είναι, είναι χαζό να βάζουμε προϋπολογισμό που χρειάζεσαι για άσκηση και προσωπικό και να κρατάς ένα μεγάλο ποσό για μία εξάμηνη ε, περίοδο, ίσως, ε, γιατί μπορεί ίσως να χρειαστεί για την ε, ομάδα αυτή. Και αν δεν αναπτύξεις την ομάδα, χάνεις τα χρήματα. Έτσι λοιπόν το χρησιμοποιούν για όλες τις άλλες δράσεις και αυτό παραμένει πρόβλημα και ελπίζω να το λύσουμε. Υποστηρίζω πλήρες τις χώρες που, που το υποστηρίζουν και είναι μόνο μία-δύο που δεν το κάνουν. Θα προσπαθήσουμε και πάλι. Ελπίζω όλοι να κατανοούν το σημαντικό λόγο που πρέπει να υπάρξει αυτή η βελτίωση. Αυτό για την Αθηνά και τις ομάδες Β. Κάθε φορά ε, λέγεται ότι πρέπει να υπάρχει μόνο μία ομάδα Β. Καταλαβαίνω το λόγο ε, να μην υπάρξει αύξηση σε διάφορους τομείς, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλους οργανισμούς ε, όπως ο ΝΑΤΟ, το υποστηρίζω πλήρως. Ήταν σημαντικό να γίνει αύξηση των δυνατοτήτων σε άλλους τομείς, ας πούμε το Αφγανιστάν. Σε αυτή την περίπτωση απλώς αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν προτεραιότητες. Και είναι δύσκολο σε αυτή την περίοδο να έχουμε όλες τις ομάδες Όμως ε, η αρχική ιδέα είναι ότι ε, τα χρειαζόμαστε αυτά, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το μηχανισμό. Τώρα, η συγκέντρωση και το διαχωρισμός ε, των ε, κριτηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ε, νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να διευκολύνουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ή να πάνε στον ΝΑΤΟ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο όφελος. και αυτό δεν έχει να κάνει με αυτά που κάνω εγώ, γιατί κάνω λίγο πολύ αυτά που κάνει μια στρατιωτική επιτροπή στο ΝΑΤΟ, αλλά έχουμε και άλλες χώρες Οπότε μπορούμε να βρούμε συνέργειες με αυτές τις χώρες και να υπάρχει στενός συντονισμός με το ΝΑΤΟ για να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Όμως το όφελος ε, της χρήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Αυτοί έχουν έναν μικρό προϋπολογισμό, αλλά έχουν προϋπολογισμό για την τεχνολογία και την ανάπτυξη. Αν είναι χρήσιμος, μπορεί ας πούμε, ένα μέρος του να συνδεθεί με τα δικά σας project. Και είναι σημαντικό ότι ο ΕΟΑ έχει ε, στο είναι εντολή του την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε ε, ισχυρό στρατό, θέλουμε ισχυρή οικονομία ταυτόχρονα. Και νομίζω ότι γι' αυτό το, δρο... το λόγο είναι χρήσιμο αυτό να το λάβουμε υπόψη μας, μεταξύ άλλων. Ε, υπάρχουν επίσης και άλλα ε, θέματα που θέτουν τα κράτη. Ε, γιατί να ζητάμε ICT αν θέλουμε κάτι γρήγορα ε, και δεν υπάρχει τεχνολογία και πρέπει να την αναπτύξουμε, θα χρειαστεί χρόνο. Αν τη χρειαζόμαστε γρήγορα, μπορεί να πάμε σε έναν εταίρο που μπορεί να μας βοηθήσει γρήγορα και να περάσουμε μέσα από το ICT που έχει ε, Συνδέσμος με την διοίκηση των δυνάμεων και αυτό με την βιομηχανία. Και οι ευρωπαϊκέ και οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες όλες έχουν ε, σχέσεις και συνδέσμους. Ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους αποδοτικούς τρόπους που υπάρχουν για να έχουμε τις κατάλληλες ε, υποδομέ και ικανότητε. Τώρα για τη χαμηλή πολιτική βούληση νομίζω ότι την κάλυψα έχει να κάνει με την ε, οικονομική κρίση. Μετά είπαμε πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα της κρίσης. Αρχικά ε, δεν έγινε οργανωμένη προσπάθεια. Ο κύριος Μιωτό έκανε μια καλή δουλειά με τη δική του εμπειρία και περιέγραψε τις διαδικασίες. Και έτσι αποκαλέσαμε αυτό πλατφόρμα κρίσης. Έτσι λοιπόν έχουμε το Συμβούλιο Διαχείρισης της Κρίσεως, όπου όλοι οι διαφορετικοί παίκτες που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι σε επίπεδο πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων από την Κομισιόν τουλάχιστον, έχουμε και την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ για τις ανθρωπιστικές δράσεις και τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ για το συντονισμό και όλες τις μορφές ε, ανάπτυξης ε, έργων ε, συντονισμού στο θέατρο των επιχειρήσεων και συναντηθήκαμε, αναλύσαμε την κρίση. Μία από τις ερωτήσεις είχε να κάνει με τις, με τις πληροφορίες ασφαλείας. Υπήρχε μια τέτοια ερώτηση για το κέντρο επιχειρήσεων. Από τη δική μου πλευρά τη στρατιωτική να πω ότι συνεργάζονται στενά, βρίσκονται στον ίδιο, στο ίδιο κτίριο, όχι σε δύο διαφορετικούς οργανισμούς. Γεωγραφικά και μη λοιπόν είναι κοντά και συνεργάζονται με κοινά έγγραφα κτλ. Άρα η κατάσταση ε, στην ουσία έχει να κάνει με μια μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της πλατφόρμας ε, κρίσεων και υπάρχει το Situation Center που είναι το, έχει την αίθουσα SIT που είναι εκεί που υπάρχουν οι πληροφορίες και είναι μια δυνατότητα που με την πρωτοβουλία του κύριου Μιότζο μπόρεσε να συγκεντρώσει και τα 27 κομμάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από την εξωτερική υπηρεσία. 24 ε, ώρες το 24ωρο και κάθε μέρα της εβδομάδας. Έχουμε λοιπόν ε, δύο ωφέλη. Γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, χρησιμοποιούμε το προσωπικό. Πάντοτε μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο και κάποιος είναι εκεί και βελτιώνει την ποιότητα των πληροφοριών. Οι δικοί μου άνθρωποι που κάνουν εκθέσεις για τις αποστολές, αναφέρονται για τις αποστολές, λέμε ας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια ε, δράση εναντίον της πειρατείας και την διέκοψε. Μπορεί να έχουμε και το ΝΑΤΟ που να εμπλέκεται. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικούς ανθρώπους που κάθονται ένας απέναντι στον άλλον. Ελέγχουμε ποια είναι η αλήθεια και η πραγματική ιστορία πηγαίνει στην οικεσία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβετε λίγο πολύ ε, πώς έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, το Citroom είναι οι καθημερινέ πληροφορίε που συγκεντρώνονται από τι επιχειρήσει ανοιχτέ πηγέ και υπάρχει και ένας ε, ε, σύνδεσμος με τις πληροφορίες ασφαλείας για να ελεγχθεί αν υπάρχουν πληροφορίες που δεν είναι σωστές. Αυτή είναι η κατάσταση για την συλλογή πληροφοριών και τη διοχέτευση στην ηγεσία. Τώρα, να μην ξεχνάμε την αλλαγή του κλίματος. Το, η αλλαγή του κλίματος είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όχι που μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς για αυτό το θέμα, αλλά με τη δική μας ανάλυση, νομίζω πως μπορεί, όταν μιλάμε για ασφάλεια, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επί της ασφάλειας και της ασφάλειας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν μακροχρόνια για να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύσσουμε μια στρατηγική η οποία μπορεί να βοηθήσει αυτό ποιες είναι εκείνες οι απαραίτητες τεχνολογίες και τις ανάγκες που θα έχουμε, ε, πόσον προβάλλουμε αυτό το σχήμα στο μέλλον και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις επίσης αυτής της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι, ε, της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι προφανές. Και τι αυτό σημαίνει ενδεχομένω 5-10 χρόνια, επόμενα 5-10, κατά πόσον η θαλάσσιοι ότι θα είναι ανοιχτή στον Καναδά για παράδειγμα, στην Ευρασία και το κατάλληλο. Βεβαίω, σε αυτή την αλλαγή πρέπει να έχουμε μια στρατηγική, σε ένα στρατηγικό σκεπτικό. Και αυτό πρέπει και στην Αφρική να ισχύσει, αλλά ακόμη και στον πάγο μπορεί να υπάρχουν λύσεις, ιδιαίτερα όταν δει πραγματικά κανένα ότι μπορεί να υπάρξει μια άνοδος της στάθμης των υδάτων Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα στρατηγικό θέμα και θα πρέπει να ειδωθεί, να ειδωθεί και να ληφθεί υπόψη γενικότερα σε αυτή τη στρατηγική της αλλαγής του κλίματος του προσωπικού, του επιτελείου, ποια θα είναι η ποιότητα. Αυτό έθεσε σαν ερώτημα προηγουμένω. Υπάρχει ένα σχεδιασμός και όλα αυτά τα μέλη βεβαίως που θα υπάρχουν στο προσωπικό του επιτελείου έρχονται από τα κράτη-μέλη και, και βεβαίως υπάρχουν οι παροχέ οι οποίες προβλέπονται, οι πληρωμέ οι οποίες υπάρχουν για αυτό το προσωπικό, καθώς επίσης και τα κονδύλια εκείνα ένα άτομα του, αυτού του συνδύματος είναι αυτή τη στιγμή το μη στρατιωτικό προσωπικό. Κάθε τρία χρόνια το προσλαμβάνουμε και αυτό το κάνουμε σε κάθε σύστημα, παντού. Όλοι ξεκινάνε από το χαμηλότερο επίπεδο και φεύγουν βέβαια στο ψηλότερο. Και ξέρετε αυτό το πυραμιδικό τι σημαίνει ότι σιγά σιγά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα προλαμβάνει κάθε τρία χρόνια νέο προσωπικό, μη στρατιωτικό, βεβαίως ότι υπάρχουν δυσκολίες και ότι θα πρέπει κάθε τρία χρόνια να αλλάζει το 1 τρίτο του προσωπικού το οποίο ασχολείται με αυτό το θέμα. Και αυτό καταλαβαίνε. Είμαστε πολλοί νέοι, ιδιαίτερα οι νέοι είναι το στρατιωτικό προσωπικό και όλες οι διαδικασίες οι οποίες για τους στρατιωτικούς σε ε, στρατιωτικό πρόγραμμα λειτουργικό, επιχειρησιακό η, για όλες τις χώρες και όλα τα επίπεδα το σύστημα είναι το ίδιο, είναι συνολικό, είναι πλήρες και καλύπτει όλο, το, όλο αυτό το προσωπικό από ανεξαρτήτως χώρες από την οποία προέρχονται οι στρατιωτικοί ή μη στρατιωτικοί. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως η συνάδελφος ήθελε να παρέμει και να θέσει ένα ερώτημα παρακαλώ ίσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ερώτηση. Μετά τη Λιβύη, Λιβύη έγιναν πολλά πολλέ συζητήσει όσον αφορά τι ικανότητε τη ΕΕ και τη Ευρώπη, πώ μπορεί να κάνει και τι έπρεπε να κάνει. Ποια είναι τα μαθήματα, τα πορίσματα, τα διδάγματα, αν θέλετε, και κατά πόσον μια τέτοια ίδια επιχείρηση μπορεί να γίνει στα πλαίσια της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Δεύτερο, όσον αφορά τις ομάδες επιχειρησιακής, ε, τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εμπόλεμες. Αυτές χρειάζονται χρήμα. Ξέρετε ότι είμαστε εγώ στην κυβέρνηση της χώρας μου, της Φιλανδίας, όταν έγινε αυτή η συζήτηση και κατά πόσον αυτοί οι επιχειρησιακές εμπόλεμες ε, θα πρέπει να έχουν χρήματα διότι είναι παρούσες εκεί. Και αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Βεβαίω καλύτερα θα ήταν να μην χρησιμοποιούνται, αχρίαστε να είναι θα λέγαμε στα ελληνικά. Αλλά όταν χρειαστούν, ε, πρέπει, χρειάζεται και χρήμα το οποίο θα πρέπει να πέσει επί της τραπέζης. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω πως σε τέτοιου είδους καταστάσει χρειάζεται χρήμα. Ευχαριστώ επί του θέματο αξίζει το πρώτο ερώτημά σα θα χρειαστεί μια ολόκληρη ακρόαση όσον αφορά τη Λιβύη και τα κατοπινά την επόμενη μέρα της Λιβύης. Παρακαλώ στρατηγέ μου, μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μου δίνετε η ευκαιρία να πω δύο πράγματα για τη Λιβύη. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα τα οποία τα επεξεργαζόμαστε σε επίπεδο τακτικής αλλά, ε, της χώρας μέλη και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Αυτή η συνήθιση διαδικασία για οτιδήποτε κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μία αρκετά επιτυχή εμπλοκή στην Ένωση των ε, Ευρωπαίων πολιτών ε, από τη Λιβύη. Ήμασταν μέρος του μηχανισμού αυτού εκένωσης. Όλα αυτά αποφασίστηκαν ε, σε μια συντονισμένη ομάδα. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση μπορέσαμε να δώσουμε τις πληροφορίες εκεί που ήταν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημερώθηκε το προσωπικό μου που επικοινωνεί με όλα τα Υπουργεία Άμυνας, συγκεντρώθηκαν όλες οι πληροφορίες και με αυτόν τον τρόπο εκενώθηκαν ε, πάρα πολύ, έγινε και ένωση πολλών αμάχων. Μάθαμε πάρα πολλά από αυτό το μηχανισμό. Απεδείχθη ότι ήταν ιδιαίτερα καλός. Σε στενή συνεργασία με την ΕΚΟ υποστηρίξαμε, στηρίξαμε τους πρόσφυγες από την, ε, την Ισία όταν ο ρυθμός τους έγινε ιδιαίτερα υψηλός και δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες υποδομές. Οφεληθήκαμε πολύ από αυτό. Μόλις βρω μια χώρα μέλος που είναι διατεθειμένη να αναλάβει τη μεταφορά, τίθεται σε διαδικασία. Είναι η διαδικασία που περατώνται μέσα σε 24 ώρες. Δείξατε και ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα στο ΜΕΑΣ όπου έμαθε περισσότερα το ΝΑΤΟ. Έδωσε τέλος σε μία επέμβαση και το θέμα είναι ότι η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει μόνη της. Χρειαζόμασταν την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, χρειαζόμασταν τις υποδομές που έχουν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτή βεβαίως είναι μια δυναμία. Αν θέλουμε να επιτευχθεί ο στόχος μας και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωση, πέρα από το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθεια, φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένας λόγος ύπαρξης για τους στρατιωτικούς ε, να εργάζονται από κοινού, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέχρι το επίπεδο που μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή την ε, εδραίωση της ειρήνης. Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται ξεχωριστές ομάδες, ε, θα πρέπει να διαχωριστούν ομάδες που, που είναι αντικρουόμενες. Χρειάζονται αυτές οι υποδομές τα μαθήματα που μάθαμε από το ΝΑΤΟ είναι πολλά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για μας, γιατί θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε την βεβαιότητα ότι έχουμε τις υποδομές πιο περιορισμένες της Ατλαντικής ε, Συμμαχίας, αλλά που μας επιτρέπουν ε, να φέρουμε εις πέρας πολύπλοκες στρατιωτικές ε, δράσεις. Είδα ότι στην ε, έκθεση έγινε μια αναφορά στον προπολογισμό για τις αποστολές και την τεχνολογία. Βεβαίως οι προπολογισμοί έχουν συρρυκνωθεί σε όλες τις χώρες και αν θέλουμε να επενδύσουμε σε νέες υποδομές, γιατί για τις περισσότερες χώρες ε, μέλη ε, μιλάμε για νέες υποδομές, θα πρέπει να γίνουν περικοπές σε πολλά επίπεδα υποδομών και μετά θα πρέπει να υποβάλουμε το αίτημα να συρρικνωθούν ακόμα περισσότερο αυτές οι υποδομές και ο, να δοθεί ένας προϋπολογισμός στην ε, Ευρωπαϊκή, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Άμυνα, στην DDA. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το κάνουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ο χειρότερο, η χειρότερη στιγμή για να θέσουμε ένα τέτοιο ερώτημα. Και βλέπετε λοιπόν λοιπόν ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτά τα κοινά τεχνολογικά προγράμματα. Για μένα δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι ουσιώδες το πρόβλημα. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Παρακαλώ και Στατιέ. Η ομάδα μάχης Πήραμε το παράδειγμα της Φιλανδίας. Φιλανδία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η Φιλανδία ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτή την ομάδα μάχης σε ένα πλαίσιο που ήταν ε, καλό, το Τσάντ. Διεξήχθη μια δημόσια συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Μόλις υπάρχει όμως μια χώρα μέλος που δεν συμφωνεί με την κρίση του, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ούτε η Φιλανδία δεν, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι φιλανδικές υποδομές ε, ε, στο Τσάντ. Συνεπώς η ε, δαπάνη που κινούν είναι πολύ σημαντική. Μπορώ να παραθέσω πολλά παραδείγματα επί των ημερών μου, δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε βελτιώσει τον προγραμματισμό. Και υπήρξαν σενάρια όπου μια καλύτερη ομάδα θα ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα υποστήριζε ε, θα ήταν υποστηρικτικό μηχανισμό στην εκένωση ε, ή στην παρουσία υποστήριξη ή ε, στην αύξηση των υποδομών. Βεβαίω η ομάδα αυτή, η καλλιτέχνη ομάδα είναι ένα η πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά ελπίζω ότι θα επιτευχθεί η συνένεση τελικά έτσι ώστε μεταξύ των άλλων να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τον, ε, το χρηματοπιστωτικό μηχανισμό. Δεν είναι μόνον αυτός, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για πολλές χώρες μέλη. Ευχαριστώ στρατηγέ, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που κάνετε, ευχαριστώ που ήσασταν διαθέσιμος. Ο πρέσβη κύριο Στίβεν, θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συντοδομία. Βεβαίω το Αταλάντα Foster είναι πρόβλημα για την Αταλάντα, αλλά και για την ε, Βοσνία, αλλά και για το Κοσυφοπέδιο, Και εκεί έχουμε πρόβλημα, στο βόρειο Κόσοβο, Αταλάντα. Εκεί χρειάζεται ένας ελάχιστος αριθμός αναγνωριστικών σκαφών και ε, σκαφών υπήρχε, αντιμετωπίσαμε πρόβλημα τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τους υπόλοιπους μήνες δεν υπήρχε πρόβλημα. Ένα, ένα στοιχείο, ένα στοιχείο. Το γεγονός ότι είχαμε προβλήματα αποτέλεσε έναυσμα για να σκεφτούμε ε, οι ε, Ρώσοι, οι Κινέζοι κινητοποιήθηκαν ε, είπαν ότι θα μπορούσαν να, δώσουν ε, πετρελαιοφόρα. Οι Ινδοί και εκείνοι το Δεκέμβριο είπαν ότι θα αναλάβουν ορισμένα καθήκοντα στον τομέα του αυτό. Βεβαίω ε, χρειάζεται μια περισσότερο συνετή χρήση των υποδομών. Να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική προστασία των σκαφών από την ε, ε πειρατεία. Ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να, δώσει, να παράσχει άτομα τα οποία θα εκπαιδεύσουμε ε, εμείς. Αυτό κάνουμε τώρα. Προσπαθούμε να βρούμε νέες τεχνικές για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την όλη προσέγγιση μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στρατηγέ, κύριε Πρέσβη. Δίχως άλλο, μετά την ενεργοποίηση αυτού του κέντρου θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά στις τρεις αυτές αποστολές, οι οποίες ελπίζουμε ότι έχουν καλού συντονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσουμε και πάλι στις τρεις. Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα μιλήσει ο ειδικό απεσταλμένος το κέρας της Αφρικής.